στην Τινησία. Και καλό την εισηγήτρια να πάρει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους ε, που ε, ε, έπαιξαν πολύ το ρόλο τους, έκαναν πολλή δουλειά για την απόφαση που θα πάρουμε γιατί ξέρουμε ότι είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία για την Τινησία και πρέπει να σταθούμε στο πλευρό της. Όλοι γνωρίζετε τις προκλήσεις, ε, τις τόσο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει την Ισία, οικονομικές προκλήσεις, ανεργία που έχει εκθετική ανάπτυξη, τρομερές ε, περιφερειακές ανισότητες μεταξύ της Τίνιδας και της υπόλοιπης ισίας, οικονομικές προκλήσεις, γιατί φυσικά όλοι θυμόμαστε τις τρομοκρατικές επιθέσεις που διέλυσαν τον τουρισμό από τον οποίο εξαρτώνται 500.000 θέσει εργασία. Και σήμερα δεν υπάρχει τουρισμός στην την προβλήματα ασφαλείας. Αν οι συνάδελφοι μπορούσαν ε, να ησυχάσουν θα μπορούσα να συνεχίσω την ομιλία μου. Προκλήσεις λοιπόν για την ασφάλεια. Θυμόμαστε όλοι την τρομοκρατική επίθεση στο Μουσείο Μπαρντό και στο ΣΟΥΣ. Ε, θυμόμαστε τι έγινε και στα σύνορα την Ισίας Λιβύης η Τινησία έχει περίπου 500 χιλιόμετρα συνόρων με τη Λιβύη που είναι απόλυτα αποσταθεροποιημένη με όλες τις διακινήσεις ε, ανθρωπίνων, ε, όντων, ναρκωτικών, ε, τα προβλήματα της τρομοκρατίας και θυμίζω ότι οι φίλοι μας οι Τινήσοι φιλοξενούν 1,8 εκατομμύρια προσφύγων από τη Λιβύη που είναι περίπου 20% του πληθυσμού. Να λοιπόν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η Τινήση και παρά τις προκλήσεις αυτές η Τινησία ανταποκρίνεται είναι δημοκρατική χώρα η δημοκρατική μετάβαση είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη και η κοινωνία των πολιτών στην ε, Τινησία έλαβε βραβείο Νόμπελ για να ενθαρρυνθούν αυτές οι προσπάθειες και παρά το ότι επιμένει σε αντίξω συνθήκε στην πορεία τη η Τινησία σημαίνει ότι πρέπει να τη συμπαρασταθούμε και γι' αυτό υποβάλλουμε αυτό το πρόγραμμα 500 εκατομμυρίων μακροοικονομική συνδρομή στην Τινησία. Χρειάζεται αυτό το κεφάλαιο η Τινησία. Το σχέδιο αυτό εντάσσεται στα πλαίσια τη στρατηγική μα γενικά για την Τινησία. Έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσει, οι εμπορικέ διαπραγματεύσει και θα επιθυμούσα να τονίσω ότι συζητάμε στην ουσία μια εταιρική σχέση πολιτική και οικονομική με αυτή τη χώρα. Έχουμε λάβει τα αναγκαία επίγοντα μέτρα με τις ποσοστώσεις 35.000 ε, τόνοι ετησίως ε, χωρίς δασμούς και σήμερα συζητούμε αυτήν την ε, μακροοικονομική χρηματοδοτική, την δεύτερη για 15 χρόνια που εξαρτάται από ορισμένε μεταρρυθμίσεις που θα ήθελα όντως να είναι οι κατάλληλες να μην είναι απλώς λογιστικές, να βοηθήσουν λοιπόν ουσιοδό στην ανάπτυξη της χώρας. Εάν εγκριθεί αυτή η έκθεση, κάτι που ελπίζω να συμβεί ε, σε λίγο, πιστεύω ότι και το Συμβούλιο θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια και καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τις εκταμιεύσεις αυτών των κεφαλαίων τάχιστα, πριν το καλοκαίρι, πριν τις διακοπές δηλαδή, γιατί χρειάζεται τα κεφάλαια αυτά η Τινησία. Αυτή η συνδρομή ορισμένοι μπορούν να θεωρούν ότι είναι απλώς μια επιδότηση όχι, δεν είναι επιδότηση, είναι δάνειο που θα πρέπει να επιστραφεί. Και θέλω να μιλήσω και για το όλο και αυξανόμενο χρέος της Τινησίας και θέλω να το συζητήσουμε αυτό. Χαίρομαι που μας ακούει εδώ η Επιτροπή και η Γαλλία και η Γερμανία αποφάσισαν ένα τμήμα του χρέους, τους, ε, του χρέους της Τινησίας έναντι αυτών 60 εκατομμύρια και για τη Γαλλία και τη Γερμανία αποφάσισαν λοιπόν να μετατραπεί αυτό το χρέος σε ε, χρηματοδότηση ανάπτυξης της Τινησία. Νομίζω ότι είναι σωστή και ευφύη λύση και καλό την Επιτροπή στο μέλλον, πέρα από το σχέδιο που θα εγκρίνουμε τώρα, να εξετάσει κάποια παρόμοια προσέγγιση θα ήταν πιο χρήσιμο, πιο σκόπιμο για την Τινησία αυτό που έκανε η Γαλλία και η Γερμανία να το μιμηθούν. Νομίζω πως θα μπορούσε να προτείνει η Κομισιόν τέτοιες πρωτοβουλίες. Ξέρουμε όλοι λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε στο πλευρό της Τινησίας και των κατοίκων της όχι μόνο προ οφελό του, αλλά και προ το δικό μας όφελος. Χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μια σταθερή, ειρηνική και ευημερούσα την Ισία. Πρέπει να είμαστε στο πλευρό της. Σας ευχαριστώ όλου. Ευχαριστώ. Ο επίτροπο Κατάινα. Αξιότιμη. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω την κυρία Ντεσαρνέ, καθώ επίση και την Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου για την έκθεση αυτή. Όπω ξέρετε, και όπω ξέρουμε όλοι, η Τινησία αντιμετωπίζει πολύ σημαντικέ οικονομικέ προκλήσει και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε την πρόταση αυτή για μακροοικονομική συνδρομή προ την Τινησία. Η Τινησία λοιπόν αντιμετωπίζει τι συνέπειε των τρομοκρατικών επιθέσεων του 2015. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο κλάδος του τουρισμού, ιδίω ο κλάδος του τουρισμού, έχει πειραστεί ιδιαίτερα δεινά και οι ξένες επενδύσεις έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε πολύ μικρή άφηξη ξένου συναλλαγματός και ξένων επενδύσεων στη χώρα αυτή. Χρειάζεται λοιπόν τη μακροοικονομική αυτή συνδρομή η Ισία προκειμένου να καταφέρει να σταθεροποιηθεί και προκειμένου να συνεχιστεί η δημοκρατική της μετάβαση η οποία ξεκίνησε μετά την Αραβική Άνοιξη. Στην ε, διάσκεψη των δωρητών επικεφαλής του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατέστη σαφέ ότι πρέπει να υποστηρίξουμε χρηματοοικονομικά την Ισία και τώρα και στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πρέπει να συμβάλλει στην ε, ανανεωμένη αυτή μακροοικονομική συνδρομή προς την Ισία και το προτείνουμε αυτό δίνοντας μια νέα τέτοια υποστήριξη 500 εκατομμυρίων ευρώ. Μια υποστήριξη η οποία βασίζεται στην προηγούμενη συνδρομή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με 300 εκατομμύρια ευρώ. Προβλέπετε λοιπόν ότι η νέα αυτή χρηματοοικονομική συνδρομή, η νέα αυτή υποστήριξη που είναι το μεγαλύτερο τέτοιο ποσό που δίνεται προς τη χώρα αυτή και προς τις χώρες της νοτίας γειτονίας εν γέννη, θα δοθεί μέσω τριών δόσεων τα επόμενα τρία χρόνια. Η εξαιρετική λοιπόν αυτή έκτακτη συνδρομή που δίνεται στην Τινησία θα πρέπει να ειδωθεί και στα πλαίσια του γενικότερου πλαισίου προόδου που έχει σημειώσει την Ισία τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να καταφέρει να έχει ένα καλός ένα σύστημα δημοκρατικό το οποίο θα λειτουργεί ομαλά και αποτελεσματικά. Η νέα αυτή χρηματοοικονομική συνδρομή βέβαια θα βασίζεται σε διάφορες πολιτικές προϋποθέσεις. Όντως η Τινησία θα πρέπει να εφαρμόσει τα νέα προγράμματα του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου και όλες τις οικονομικές και πολιτικές προϋποθέσεις σχετικές προκειμένου να ικανοποιήσει όλες τις αιτήσεις που υπάρχουν στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεννόησης. Καλύπτονται πάρα πολλοί τομείς όπως η φορολογική μεταρρύθμιση, η ενίσχυση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν προκειμένου να αποκατασταθεί ο τουρισμός, το εμπόριο και οι υπηρεσίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Ο χρόνος πιέζει. Είναι πολύ σημαντικό μέσω της μακροοικονομικής αυτής συνδρομής να καλυφθούν οι εξωτερικές οικονομικές ανάγκες της ε, Τινησίας για το 2016 και το 2017. Πρέπει λοιπόν να εγκρίνουμε όσοι νομοθέτες το συντομότερο δυνατό τη νέα αυτή πρόταση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο χαίρομαι ιδιαίτερα που η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου ενέκρινε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρί τροπολογίε. Χαίρομαι επίση πάρα πολύ που το Συμβούλιο στην επιστολή στα πλαίσια τη Κορεπέρα είπε ότι πρόκειται να υποστηρίξει την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρί περαιτέρω τροποποιήσει αφού βέβαια εγκριθεί πρώτα η πρόταση αυτή και από εσά σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα και προσβλέπω σε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και τώρα αρχίζει ο κατάλογος των ομιλητών για 1,5 λεπτό ο κύριος Τσίκου. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε εξ ονόματος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Υποστηρίζω πολύ στεναρά την πρόταση αυτή. Νομίζω πραγματικά ότι επίγει η οικονομική αυτή υποστήριξη προς την Ισία για όλους αυτούς τους λόγους που ακούσαμε. Ας αναφερθώ λίγο στους λόγους αυτούς. Καταρχάς, η πολιτική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια πολιτική πάρα πολύ σημαντική, ένα πολύ σημαντικό και αποτελεσματικό μέσο, καθότι βασίζεται σε ένα δημοκρατικό σχέδιο, σε ένα σχέδιο εδραίωσης τη δημοκρατία και τη ελευθερία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να προωθήσουμε το σχέδιο αυτό της πολιτικής γειτονία και προ τα νότια της Ευρώπης. Και είναι πολύ σημαντικό να τηρούνται συγκεκριμένε προποθέσει και να λάβουμε υπόψη μας και το πρόβλημα της προσφυγικής κρίσης, το οποίο επιδεινώνει την κατάσταση και πολλές φορές μας κάνει να αναβάλουμε κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Πιστεύω ότι τώρα θα πρέπει να επικεντρωθούμε ακριβώς σε αποτελεσματικές πολιτικές. Από την άλλη υπάρχει και το πρόβλημα των διαθροτικών μεταρρυθμίσεων που πρέπει να κάνει την Ισία. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα αντιστοιχούσαν σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 500 εκατομμύρια ευρώ που προτιθέμεθα εμείς να δώσουμε είναι μια σημαντική συμβολή προκειμένου να κινηθεί η Τινησία προς σωστό δρόμο. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα λοιπόν υποστηρίζει την πρόταση αυτή, δεν υπέβαλε τροπολογίες, είναι όμως σαφές ότι ε, είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούνται πάντα οι κανόνες και οι βασικές προϋποθέσεις και είναι πολύ σημαντικό στο όνομα του γενικού και ευρωπαϊκού συμφέροντος αλλά και στο όνομα του συμφέροντος της Τινησίας είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κύριος Μορέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από την εποχή που ξεκίνησαν οι τινήσοι την πορεία για τη δημοκρατική μετάβαση, όλοι εδώ θυμόμαστε την υποδειγματική του στάση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε στάθηκε αλληλέγγυο προς την Τινησία και τους Τινήσιους. Ε, ξεκινήσαμε μια διαδικασία ε, συμφωνίας ελεύθερων ανταλλαγών. Φυσικά ε, ξέραμε ότι αυτό είναι μια ασύμετρη και προοδευτική εταιρική σχέση με την Τινησία και βεβαίως όταν χρειάστηκε να μειώσουμε την ποσόστοση για το ελαιόλαδο της ε, την Ισία φτάσαμε σήμερα στο θέμα της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής προς την, ε, την Ισία. Είναι κατεπήγον το θέμα και γι' αυτό το λόγο είμαστε υπέρ. Αλλά υπάρχουν και διάφορα που πρέπει να θυμηθούμε στη συζήτηση αυτή. Πρώτον, όταν λέμε ότι η Τινησία πρέπει να είναι σε θέση να κάνει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Καλό την Κομισιόν να υπάρξει ευέλικτη, ευφυής απέναντι σε αυτό, γιατί δεν θέλουμε να πνίξουμε εντελώς την οικονομία της χώρας. Δεύτερον, μιλάμε για το δουνουτού, αλλά αυτό σημαίνει δάνεια. Δάνεια σημαίνει χρέο αλλά το, το χρέος της Ινησίας σήμερα αποτελεί πρόβλημα το οποίο κληροδοτήθηκε από την περίοδο Μπεναλή. Δεν πρέπει λοιπόν τα χρήματα που ε, δανείζουμε στην Τινησία να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αποπληρωμή του χρέους του προηγούμενου καθεστώτος. Άλλο πολύ σημαντικό για μας πρόβλημα. Υπάρχουν πολλοί υποδοί του Μπεναλή στην Ευρώπη και βεβαίως πρέπει να γίνει από... Ε, ε, πλευράς Ευρώπης για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Αν είμαστε υπέρ αυτής της κατεπίγουσας βοήθειας ξέρουμε ταυτόχρονα ότι μακροπρόθεσμα πρέπει να έχουμε σταθερή αλληλεγγύη και να μην ε, χρησιμοποιούμε μόνο τις κατεπίγουσες ενισχύσεις. Και γι' αυτό το λόγο εμείς σοσιαλδημοκράτες είμαστε υπέρ. Ευχαριστώ κύριος Λούνατς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, χαιρετίζω τους καλεσμένους στα θεωρία. Ε, η Ευρώπη πρέπει να κοιτάξει τις τεράστιες ευθύνες και τις δυσκολίες που έχουμε. Η Τινησία σταθεροποιείται ξαναδημιουργεί την δημοκρατία και αναδύεται από μία περίοδο τεράστιων οικονομικών και πολιτικών ε, δυσκολιών. Υπάρχει υψηλή ανεργία των νέων, θέματα ασφάλειας, τρομοκρατίας και αυτή, αυτού του είδους η βοήθεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Η Τινησία πρέπει να είναι αξιόπιστος και σταθερός εταίρος στην περιοχή. Πρέπει λοιπόν να της προσφέρουμε υποστήριξη σε αυτή τη δύσκολη μετάβαση προς την δημοκρατική σταθερότητα πολιτική αυτή είναι κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Δίνουμε οικονομική ενίσχυση στην περιοχή αυτή. Μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξή μας, αλλά δεν δίνουμε λευκή επιταγή. Περιμένουμε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις που θα δημιουργήσουν ε, θέσεις εργασίας. Ένα λεπτό για τον κύριο Λεό. Ευχαριστώ. Πρέπει να βοηθήσουμε τους τρινήσιους. Πρέπει να τονίσουμε ότι επιδεικνύει τρομερή υπευθυνότητα η κοινωνία, οι συνδικαλιστικές ενώσεις, οι πολιτικές δυνάμεις για να συνεχιστούν οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και να βελτιωθεί η ζωή των τυνησίων. Αλλά η βοήθεια αυτή δεν μπορεί να γίνει με τις παλιές αντιλήψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που αυξάνουν το χρέος και μειώνουν την λαϊκή κυριαρχία. Πρέπει να βοηθήσουμε την Τινησία και γενικότερα με τους λαούς του Νότου με τρόπο πιο τολμηρό, πιο εφευρετικό για να δημιουργήσουμε ε, ενός είδους, ε, μία ενός είδους κοινή τράπεζα, κοινό ταμείο για να παγώσουν ε, τα χρέη και να δημιουργήσουμε διαρκή ανάπτυξη που να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και την ανθρώπινη και οικολογική ανάπτυξη. Και είναι επιτέλους χρόνος να επιστραφούν τα περιουσιακά στοιχεία που είχε το καθεστώς Μπεναλή και να δοθούν πίσω στο λαό. Δύο λεπτά ο κύριος Ζαντό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ξέρουμε την κατάσταση στην Τινησία. Είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Και ο λαός αντιμετωπίζει πολλές δυσχέρειες. Ξέρουμε ότι κατέρευσαν ε, οι τουριστικές δραστηριότητες λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων. Ξέρουμε τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγές της Τινησίας και καλά κάναμε που διευκολύναμε τις εξαγωγές αυτές για το ελαιόλαδο προς την Ευρώπη Ξέρουμε πόσο ευάλωτο, πόσο ευαίσθητο είναι αυτό που επιχειρούν να κάνουν την ίση για να υπάρξει δημοκρατική μετάβαση στην Τινησία ε, σε ένα έδαφος που δεν είναι μεγαλύτερο από το Ηνωμένο Βασίλειο υποδέχονται περισσότερους ε, πρόσφυγες από όσους δέχεται όλη η Ευρώπη. Και ξέρουμε πόσο μεγάλη κίνδυνοι λοιπόν υπάρχουν ε, στην γειτονία μας. Πρέπει λοιπόν πέρα από αυτά που μας ε, ζητά το... η κυβέρνηση της Τινησίας πρέπει να δώσουμε μακροοικονομική ενίσχυση στην Τινησία και ξέρουμε και είχε ψηφίσει το 2012 το Κοινοβούλιο μια παρόμοια προσέγγιση πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το απαράδεκτο χρέος της Τινησίας που υπήρξε κατά την, ε, σε μεγάλο βαθμό δημιουργήθηκε κατά την περίοδο Μπέναλη πρέπει να μειωθεί το άχθος του χρέους οι διαθροτικές μεταρρυθμίσεις που ζητάτε αγαπητοί συνάδελφοι Κοιτάξτε πώς είναι η κατάσταση σήμερα στην Τινησία και να μην θεωρείτε ότι επειδή ε, αυτή η μακροοικονομική συνδρομή σχετίζεται με τους ε, όρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν πρέπει να βοηθήσουμε περισσότερο την Τινησία. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι, πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα, πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερες παροχές προς την Τινησία. Όταν βλέπουμε τα δις που δίνουμε στην ε, κυβέρνηση της Τουρκίας που δεν είναι καθόλου πρότυπο δημοκρατίας, γιατί να μην δώσουμε πολύ περισσότερα στην Τινησία για να της επιτρέψουμε να ενισχύσει την δημοκρατική μετάβαση με βάση ανάπτυξη που να σέβεται τους πόρους και τις δυνατότητες της νησίας. Θα ήταν λάθος να μην το κάνουμε. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Καστάλντο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουμε πόσο δεινή είναι η κατάσταση της νησίας. Μας το υπενθύμησαν και οι προαλήσαντες ανεργία, ιδιαίτερα ανεργία των νέων, η τρομοκρατία που πραγματικά έχει κάνει τον κλάδο τουρισμού να γονατίσει. 1.800.000 Λίβοι οι οποίοι έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στην Τινησία και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν ε, πάρα πολλά φαινόμενα μαύρης οικονομίας στη χώρα αυτή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το δάνειο αυτό των 500 εκατομμυρίων ευρώ δεν αρκεί. Το υποστηρίζουμε σίγουρα. Θέλαμε παράλληλα η Τινησία να υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, να δείξουμε προς αυτήν αλληλεγγύη και όχι συνθήκες λιτότητας. Δεν φτάνουν λοιπόν τα δάνεια αυτά, ακόμα και αν έχουν κάποιους ευνοϊκούς όρους, ακόμα και αν μετατρέψουμε ένα μέρος του χρέους που έχει την Ισία προς την Ευρώπη σε επενδύσεις. Δεν μπορεί να εδρεωθεί η δημοκρατία σε χώρες όπου πραγματικά ισχύουν τέτοιες συνθήκες φτώχειας και τόσο μικρή οικονομική ανάπτυξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέξουμε πάρα πολύ την Ισία για να μην έχουμε νέα προβλήματα στην όλη περιοχή. Ο κύριος Μπέ έχει το λόγο. Ισλαμική Ισλαμικές τρομοκρατικές ενέργειες, πάρα πολλές απειλές, οικονομική κρίση, άνευ προηγουμένου, κατάρρευση του τουριστικού κλάδου. Πραγματικά η κατάσταση της νησίας είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και νομίζω ότι ε, έχει περάσει πλέον ο καιρό εκείνο που χαιρόμασταν πάρα πολύ για το δημοκρατικό μοντέλο τη Τινησία, για τον λεγόμενο δημοκρατικό τη μετασχηματισμό. Εγώ όμω δεν χαίρομαι αυτή τη στιγμή με το ότι μειώνονται οι δασμοί όσον αφορά τα προϊόντα. Δεν χαίρομαι για αυτή τη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, την οποία θέλετε να δημιουργήσετε μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ισία. Θεωρώ δεν θα αποφελήσει ούτε την Τινησία ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα με εσά, θεωρώ ότι η μακροοικονομική αυτή συνδρομή δεν θα ουσιαστικά προωθήσει περισσότερο την Ισία στο να φτάσει πιο κοντά στι ευρωπαϊκέ αρχέ. Βλέπω αυτή τη στιγμή ότι περισσότερο επεμβαίνουμε εκ νέου στην Ισία δημιουργώντα πιο δεινέ συνθήκε στη χώρα αυτή, δημιουργώντα περισσότερε επισφαλεί συνθήκε και δεν νομίζω πραγματικά ότι θα πρέπει να έχουμε αυτού του είδου συνεργασία η οποία ομοιάζει τελικά με κυδαιμονία. Μια παρατεταμένη περίοδο κρίσης με εκατομμύρια πολίτε τη κάτω από το όριο τη φτώχεια χώρε να βρίσκονται σε ύφεση εδώ και χρόνια και την ανεργία να καλπάζει. έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώ θα αντιδράσουν όλοι αυτοί οι άνεργοι και οι πολίτε των χωρών του νότου όπω στην ελλάδα όταν μάθουν πω η ένωση ξοδεύει δισεκατομμύρια σε βοήθεια προ τρίτε χώρε την ώρα που τι επιβάλλονται επαχθή μνημόνια αβάσταχτη φορολογία και υποθηκεύεται ο εθνικό πλούτο και η περιουσία; γνωρίζετε πως με ένα κλάσμα των χρημάτων που χαρίζεται στην τινησία οι άστεγοι που έχουν φτάσει να κοιμούνται ακόμα και έξω από το κτίριο του ευρωκοινοβουλίου στις βρυξέλλες θα είχαν τουλάχιστον μία στέγη πάνω από το κεφάλι τους. επιπλέον είναι πρόσφατη η αδοσμολόγητη εισαγωγή ελαιολάδου από την τινησία με την οποία δεν επιτρέψατε στους ευρωπαίους αγρότες να αυξήσουν και αυτοί μια φορά τα κέρδη τους. στην ελλάδα που ήταν από τις λίγες χώρες που αυτή τη χρονιά είχε παραγωγή ελαιολάδου υψηλή ποιότητας και είχαν την ευκαιρία η παραγωγοί να δουν αυξημένο το εισόδημά τους με την υπονομευτική κίνησή σας αυτή ρίξατε την τιμή τόσο πολύ που δεν θα μπορέσουν να αποσβέσουν ούτε τα έξοδα παραγωγής τους. η ιστορία μας διδάσκει πως όποτε οι δυτικές χώρες επενέβησαν στον υπόλοιπο κόσμο το αποτέλεσμα δεν ήταν παρά χειραγώγηση και εκμετάλλευση. Το κάνετε και αυτή τη φορά φορώντα ένα δίθεν φιλάνθρωπο προσωπείο. Καλύτερο λοιπόν θα ήταν να προσπαθήσετε μήπω και κάποια από τα πολλά προβλήματα τη Ευρώπη και να αφήσετε τι τρίτε χώρε να αναπτυχθούν όπω μπορούν. Καλύτερα θα τα καταφέρουν από ότι εσεί στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φίσας, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι επισμένος ότι είναι σημαντικό να στηρίξουμε αυτή τη βοήθεια, αυτή την συμπληρωματική βοήθεια 500 εκατομμυρίων. Η Τινησία είναι προνομιακός εταίρος, στρατηγικός εταίρος της Ένωσης και εκπληρεί τις δημοκρατικές προϋποθέσεις για να ωφεληθεί από αυτή τη βοήθεια. Γιατί πραγματοποιεί οικονομικές μεταρρυθμίσεις που προκρίνονται από το ΔΝΤ είναι απαραίτητο Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει τη στήριξή της σε, αυτό, σε αυτή την ε, χώρα που μετά την κακώς ονομαζόμενη Αραβική Άνοιξη μπορεί να θεωρηθεί δημοκρατική χώρα παρά τις προσπάθειες των ριζοσπαστών Ισλαμιστών για να την αποσταθεροποιήσουν. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία με τις επιπτώσεις των τρομακρατικών επιθέσεων και την ε, αποδοχή πάνω από ένα εκατομμύριο προσφύγων από τη Λιβύη και να μην ξεχνάμε ότι 3.000 διασχίζουν τα σύνορα κάθε μέρα. Επαναλαμβάνω, σε αυτή τη συγκυρία είναι απαραίτητο να δείξουμε απόλυτη βοήθεια, απόλυτη στήριξη προς αυτή τη φιλική χώρα που χρειάζεται όλο και περισσότερο να κατοχυρώσει τη Ε, Μάρτιν, ένα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το 1995 η... την ήταν η πρώτη χώρα της, Μεσογείου που υπέγραψε ε, συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα χρειάζεται τη βοήθειά μας περισσότερο παρά από Ο κύριο Μορέλ έθεσε πολύ σωστά την κατάσταση της την Βλέπουμε τρεις φάσεις εδώ. Είναι ζωτική σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα για να συνδράμει την, την Ισία να επιστρέψουν οι πόροι. Κάποια από αυτά είναι κολλημένα σε ευρωπαϊκές τράπεζες. Απαράδεκτο. Δεύτερον, θέλουμε μια βαθιά και ολοκληρωμένη ε, εμπορική συμφωνία με την Τινησία θα πρέπει να είναι ασύμετροι. Πρέπει εμεί τι αγορέ μα να ανοίξουμε περισσότερο από ό,τι αυτέ λόγω τη επισφαλού οικονομική κατάσταση στη χώρα. Και δυστυχώ, ε, και τρίτον μάλλον, ε, ε, είναι ευπρόσδεκτη αυτή η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή. Δεν περιμένουμε όμω να δώσουμε λευκή επιταγή. Θέλουμε να υπάρξει πρόοδο στην πολυκομματική δημοκρατία και το κράτο δικαίου. Ευχαριστώ, κυρία Φορέντσα. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμεί θεωρούμε ότι είναι δίκαιο να βοηθήσουμε την Τινησία προκειμένου να βγει από τη σημαντική αυτή οικονομική κρίση την οποία διανύει, ιδίω μετά τι τρομοκρατικέ επιθέσει οι οποίε έπληξαν κέριου τομεί όπω ο τουρισμό. Αλλά ακριβώ για αυτό το λόγο καταψηφίζουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπω ήδη έχουμε πει, είμαστε κατά και των μέτρων όσον αφορά το ελαιόλαδο και του δασμού. Πρέπει να υποστηρίξουμε τον τινήσιο λαό, αλλά η υποστήριξη αυτή δεν μπορεί να έρχεται απλώ μέσω ενό μέσου όπω η μακροοικονομική συνδρομή, που ουσιαστικά ακολουθεί τι προποθέσει του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και επιβάλλει διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει στην Τινησία. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 23 ετών, ε, ετών η οικονομική και κοινωνική πολιτική που ακολουθείται στην Τινησία επιβάλλεται πάρα πολύ από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Και είδαμε ότι οδηγούμαστε μόνο σε υψηλότερα επίπεδα ανισότητα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μην προχωρούμε πλέον με τη μέθοδο αυτή. Αντίθετα, θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε το χρέο, θα πρέπει να επιστραφούν τα περιουσιακά στοιχεία που έκλεψε ο Μπεναλή πίσω στην Τινησία και θα πρέπει να ακολουθήσουμε πολιτικέ οι οποίε θα αυξήσουν την οικονομία και την απασχόληση. Όχι δάνεια που θα οδηγήσουν σε νέα δάνεια. Η κυρία Σαϊφή έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις που είδαμε στην Τινησία και οι οικονομικές δυσκολίες και της Τινησίας Μα θυμίζουν ότι η Ισία πραγματικά χρειάζεται την αλληλεγγύη τη Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο από ποτέ. Όλο και περισσότερο η χώρα αυτή προσπαθεί να οδηγηθεί σε μια στάσιμη δημοκρατική κατάσταση. Το βραβείο Νόμπελ της Ειρήνης που δόθηκε στον φόρουμ διαπολιτισμικού διαλόγου για τη δημοκρατία το καταδεικνύει αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε σιγά σιγά να οδηγηθούμε σε μια οικονομική ανάκαμψη υπέρ όλων των τιμησίων και θα καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα τη ανεργία των νέων. Ένα στου τρει πτυχιούχου είναι άνεργο. Είναι πολύ σημαντικό το συντομότερο δυνατό την Ισία να επιστρέψει σε μια οικονομική ανάπτυξη και πολιτική σταθερότητα, ιδιαίτερα ευνοϊκή για το σύνολο τη περιφέρεια. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, κύριο Παντσέρη. Ο κύριος Παντσέρη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε από τις αλλαγές που είδαμε από το 2011 μέχρι σήμερα στην νότια γειτονία και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, βλέπουμε ότι την Ισία είναι η μόνη χώρα που σημείωσε επιτυχία όσον αφορά τη δημοκρατική μετάβαση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να είναι προνομιακός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποτελέσει παράγοντα σταθεροποίηση στην περιοχή, ιδίω σε σχέση με την κρίση που βλέπουμε στη Λιβύη. Έπληξε η τρομοκρατία τον τομέα του τουρισμού και γενικότερα την οικονομία της χώρας και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε μακροοικονομική συνδρομή προς τη χώρα αυτή προκειμένου να υποστηρίξουμε και την οικονομία και την κοινωνία της. Βέβαια θα πρέπει να αναλάβει το δικό της ρόλο και την Ισία. Αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ που δίνουμε προς την, την Ισία είναι μια πολύ θετική συνδρομή. Κύριε Κατάινεν όμω, λέμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα. Όπω ακριβώ κάνουμε και για την Ουκρανία. Γνωρίζοντα ότι πολλέ φορέ ε, η πολιτική λυθιότητα των εθνικιστών οδηγεί σε πολύ δεινά αποτελέσματα. Ακριβώ γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η Τινησία, αν υποστηριχθεί σωστά από εμά, μπορεί πραγματικά να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γκάλα, λεπτό. Η εισηγήτρια παρουσίασε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Τινησία. Εγώ είμαι υπέρ της επιδίωξης ευρεία συνένεσης ε, για υποστήριξη της Τινησίας σε αυτό το σώμα. Και το κάνουμε και προς το δικό μας συμφέρον. Η χώρα έχει και τις προϋποθέσεις και τη βούληση για καλύτερη συνεργασία. Θέλουμε να βοηθήσουμε αυτή τη νέα δημοκρατία να ενισχυθεί σε κάθε επίπεδο. Για παράδειγμα, για να γίνουν και οι εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι αναγκαίο. Η στήριξη που έχουμε ήδη δώσει να βελτιώσει το πλαίσιο για εξωτερικέ επενδύσει. Αυτό είναι αποφασιστικό για το θρίαμβο τη δημοκρατία και για να δημιουργηθούν θέσει εργασία. Υπάρχει εκπαιδευμένο εργατικό προσωπικό. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσει και η δική μα οικονομία τι δυνατότητε αξιοποίηση τη θέση τη χώρα αυτή στην κεντρική Μεσόγειο. Η χώρα ε, πρέπει να κάνει συγκεκριμένα βήματα για την βελτίωση τη κατάσταση τη ε, ασφάλεια. Έχουν ήδη γίνει ορισμένα, ούτω ώστε να μπορέσουν να επανέλθουν οι πολίτε μα ω τουρίστε και έτσι να συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία θέσεων εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριος Μπαστουνάρχου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις και ο διαρκής κίνδυνος νέων επιθέσεων είναι σημαντικός παράγων που επηρεάζουν, την οικονομία όπως είπαν και όλοι οι προλαλήσαντες η χώρα έχει χάσει πάνω από το 1 τρίτο των ε, τουριστών που την επισκέπτονται αλλά κυρίως η Τινησία έχει πληγεί από την αστάθεια στην περιοχή της. Όλοι σήμερα θα συμφωνήσουμε ότι είναι η μοναδική επιτυχημένη μετάβαση προς τη δημοκρατία στην περιοχή και άρα πρέπει να βοηθήσουμε την Τινησία και τους Τινήσιους. Η Ευρώπη έχει ήδη προσφέρει ουσιαστική ε, οικονομική και, τεχνική βοήθεια θα πρέπει να ε, ε, ενισχυθεί από μια ολοκληρωμένη και πλήρη συμφωνία ε, εμπορίου που πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να είναι ασύμετρη και αυτό θα ωφελήσει την Τινησία. Πιστεύω ότι είναι για μία φορά κατεπήγον να καταβάλει η Ευρώπη όσο το δυνατόν ταχύτερα τη συνδρομή προς τη χώρα αυτή και συμφωνώ με τους προλαλήσαντες να, ότι πρέπει να ευρεθούν τα περιουσιακά στοιχεία του Μπεναλή για να επιστραφούν στους τινήσους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι ο χρόνος πιέζει. Λοιπόν, το catch the eye ως το δυνατόν ε, πιο σύντομο. Κύριο Καπούτο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Τινησία μέσα σε λίγα μόνο χρόνια κατάφερε να ενισχύσει την διαδικασία εδραίωσης της δημοκρατίας την οποία ξεκίνησε και σήμερα αποτελεί πραγματική ελπίδα στην περιοχή της Νοτίου Μεσογείου. Από οικονομική όμω πλευρά η χώρα έχει πραγματικά γονατίσει. Όλο και περισσότερο ήταν θύμα τρομοκρατικών επιθέσεων με την Ισία που πραγματικά έπληξαν κυρίω τον τομέα του τουρισμού. Κέριο τομέα αυτό για την Ισία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να βοηθήσουμε την Ισία στην δύσκολη και ευαίσθητη αυτή περίοδο την οποία διανύει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να δώσουμε την επιπλέον αυτή μακροοικονομική συνδρομή προ την Τινησία προκειμένου να εδρεωθεί η οικονομική ανάπτυξη τη χώρα και να γίνουν οι απαραίτητε μεταρρυθμίσει. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρώπη με έμπρακτο τρόπο να δείξει αποφασιστικότητα αλλά και αλληλεγγύη και να δείξει ότι πραγματικά υποστηρίζει τι χώρε εκείνε οι οποίε πρόθυσαν ένα νέο δημοκρατικό μοντέλο μετά την Αραβική Άνοιξη. Σα ευχαριστώ πολύ. Τσίτσι, για λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η Τινησία είναι χώρα που την, που την χρειαζόμαστε ως εταίρο, ως δημοκρατική χώρα της Νότιας Μεσογείου, ως υπόδειγμα επιτυχημένης μετάβασης. Για μία ακόμα φορά η Τινησία βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι και ως εκ τούτου επιχειρούμε να την ενισχύσουμε με 500 εκατομμύρια ε, ευρώ είναι κατάλληλη, είναι σωστή αυτή η κίνηση. Δεν υπάρχει εναλλακτική. δάλος θα επικρατήσει χάος στη χώρα. Άρα πιστεύω ότι η σημερινή μας απόφαση αποτελεί καλό παράδειγμα για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις χώρες που πραγματικά θέλουν να γίνουν ελεύθερες και δημοκρατικές. Υποστηρίζω την έκθεση και θα την υπερψηφίσω. Ο Είμαστε υπέρ της αρχής της διεθνούς συνεργασίας και είμαστε υπέρ της βοήθειας προς χώρες που για οποιουσδήποτε λόγους έχουν σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες. Αλλά πρέπει να είναι γνήσια συνεργασία που να σέβεται την κυριαρχία κάθε κράτους και του δικαιώματός του να χρησιμοποιήσει τους πόρους του όπως θέλει και να αξιοποιήσει όποιες πολιτικές θέλει. Πρέπει η Τινησία να μεταρρυθμίσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο και το ρυθμιστικό πλαίσιο ε, και επίσης ε, αυτά, που αυτά λοιπόν που ζητιώνται δεν είναι αυτά τα οποία θα θέλαμε εμείς, δεν είναι ειλικρινή συνεργασία. Θέλουμε να τις επιβάλλουμε ένα μοντέλο με αυτά που θέλουμε. Πλήρη αφιλευθεροποίηση της οικονομίας. Είναι μεταρρυθμίσεις που επιβάλλει και στα κράτη-μέλη της η Ένωση με τα αποτελέσματα που γνωρίζουμε. Αυτή η βοήθεια υπόκειται σε ε, προϋποθέσεις τις οποίες απορρίπτουμε και θα δημιουργήσει περισσότερες ανισότητες όπως δημιουργούνται εδώ στην Ευρώπη. Ευχαριστώ ο Επίτροπος Κατάινεν για να ε, απαντήσει. Είναι συντομία, θα υπογραμμίσω τη σημασία του κατεπήγοντος της απόφασης. Και ως εκ τούτου ελπίζω ότι θα μας στηρίξει το Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Ευχαριστώ πολύ όλους. Θεωρώ ότι έχουμε ότι συμφωνούμε επ' αυτού και πρέπει προσεκτικά να μελετήσουμε την στήριξη προς την Τινησία. Είναι θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και σταθερότητα στην περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και στο τέλος για 1,5 λεπτό η εισηγήτρια κυρία Δησαρνές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι ιδιαίτερα από το γεγονός ότι όλοι συμφώνησαν, όλοι οι συνάδελφοι έκαναν την ίδια ανάλυση. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξει πραγματική αλληλεγγύη προς την Ισία, Όλοι συμφωνούμε να απευθυνθούμε στην Κομισιόν και να πούμε ότι πραγματικά είναι κατεπήγον να δοθούν οι πόροι γιατί χρειάζεται συνδρομή την Ισία. Πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις αλλά προσεκτικά για να αντιστοιχείουν οι μεταρρυθμίσεις αυτές στο σημείο που σήμερα βρίσκεται η Τινησία. Χαίρομαι πολύ λοιπόν. Στέλνουμε ακόμα μία, ένα μήνυμα προς τους Τινήσιους σε αυτή περνάτε μια δύσκολη εβδομάδα, δεν είστε μόνοι σας, η Ευρώπη βρίσκεται δίπλα σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Ντεσαρνές.